Ε, επιπλοκές ε, να πω ότι η συμφωνία μου συμφωνεί απόλυτα με τον κύριο Σαλαφράγκα έχει γίνει συμφωνία, απλά να γίνει δηλαδή ψηφοφορία Σας ευχαριστώ πολύ Σύμφωνη κυρία Ντεκάιζερ Λοιπόν, η μερίσια διάταξη προβλέπει την ε, ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Νταφ σχετικά με την προσθήκη πρωτοκόλου για την εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία είναι σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία και τη θέτω σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Νταφ. Περνάμε στη δεύτερη έκθεση του κύριου Νταφ σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ένωσης στην τσεχική δημοκρατία ε, εξετάζουμε την πρόταση ψηφίσματος θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 1 κατά τμήματα πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα με ονομαστική ε, ψηφοφορία έναρξη παρακαλώ λήξη εγκρίνεται. θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη εγκρίνεται. συγχαρητήρια στον κύριο νταφ. η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου λοπez Ιστουριθ white και της κυρία παρβανόβα σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις. με την απλοποιημένη διαδικασία θέτω σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση έναρξη παρακαλώ. λήξη. εγκρίνεται συγχαρητήρια στους εισηγητές. η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Στάσνη σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία σε ό,τι αφορά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Ο εισηγητής, ο κύριος Στάσνη, έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Στάσνη έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει τώρα για τη συνένεσή του για την ε, τελωνιακή συνεργασία με τον Καναδά σε σχέση με θέματα που αφορούν την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Η προτινόμενη συμφωνία βασίζεται στην επέκταση του προηγούμε, της προηγούμενης συμφωνίας του 1998 όσον αφορά την αμοιβαία τελωνιακή συνεργασία και τη συνεργασία για την ε, ε, διαχείριση κινδύνου αλλά και για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Πιο συγκεκριμένα η συμφωνία μιλά για την ενίσχυση των στοιχείων που αφορούν την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων και διευκολύνουν το νόμιμο εμπόριο. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις για το προπολογισμό της Ένωσης. Εξασφαλίζει και βελτιώνει τις, σχέσεις μας με τον, τις μας σχέσεις με τον Καναδά και είναι παραπληρωματική και, και βοηθητική για την συνολική εμπορική συμφωνία την οποία διαπραγματευόμαστε και τις οποίες οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν ελπίζω σύντομα. Η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Στάτσνη. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Γκίγκολτ σχετικά με την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Θέτω πρώτα απ' όλα σε ψηφοφορία την τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται οπότε ε, η, επόμενη τροπολογία καταπίπτει. Θέλω να θέσω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρότασης της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ο εισηγητής, ο κύριος Γκίκολτ, έχει το λόγο. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, μόλις ψηφίσαμε το περιεχόμενο των αλλαγών που χρειάζονται στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για να μπορέσουμε να δώσουμε τις απαραίτητες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την Τραπεζική Ένωση την οποία ζητάμε εδώ και καιρό. Δυστυχώς κάποια κράτη-μέλη δεν είναι ακόμα έτοιμα, δεν έχουν προχωρήσει στην κύρωση και η έκθεσή μου για τις ε, αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών παραμένει βεβαίως υπό την αίρεση της έκθεσης της Μαριάν Τάισεν για την κοινή τραπεζική εποπτεία οπότε θα πρέπει η τελική νομοθετική ψηφοφορία για την έκθεσή μου πρέπει να μετατεθεί για να διατηρήσουμε τον έλεγχο της δημοκρατικής διαδικασίας στο επόμενο βήμα αυτό της ε, τραπεζικής μας ένωσης. Γι' αυτό ζητάω την αναβολή της ψηφοφορίας επί του νομοθετικού ψηφίσματος. Αναβολή της ε, ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, αναβάλλεται η τελική ψηφοφορία. Και περνάμε στην έκθεση της κυρίας Τάισεν σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Θέτω πρώτα σε ψηφοφορία την τροπολογία αριθμός 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρότασης έτσι όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η εισηγήτρια, η κυρία Τάισεν, έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ ζητάω αναβολή της ψήφισης του νομοθετικού ψηφίσματος με βάση το άρθρο 57 παράγραφος 2 του κανονισμού μας με βάση το σκεπτικό που ανέπτυξε ο κύριος Σβέν Γκίγκολτ. Και όπως είπα συζητήσαμε το θέμα αυτό χτες και σήμερα και ζητάω όπως είπα αναβολή της ψήφισης του νομοθετικού ψηφισμού. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης της κυρίας Τάισερ για αναβολή της τελικής ψηφοφορίας. Κατά. Αποχές εγκρίνεται οπότε αναβάλλεται η τελική ψηφοφορία. Και περνάμε στην έκθεση της κυρίας Ρόιτοβα σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας. Η συγγήτρια κυρία Ρόιτοβα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ κυρία Ρόιτοβα. Vážení Κύριοι συνάδελφοι, αυτή η οδηγία είναι μία από τις εννιά οδηγίες για το θέμα αυτό. Διότι αλλιώς η κατασκευή αεροσάκων σε ολόκληρη την Ευρώπη θα ήταν παράνομη από την 4η Ιουλίου. Έχουμε αλλάξει τους νόμους για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές μας καλύτερα. Ε, περιπτώσεις προϊόντων χαμηλής ποιότητας που εισάγονται στην Ευρώπη από την Ασία. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στον εξορισμό της οδηγίας. Ευχαριστώ. Και πρώτα θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 52 της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και της ομάδας του ΕΛΚ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει η επόμενη τροπολογία Θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρότασης έτσι όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και θέτω τώρα σε ψηφοφορία το σύνολο του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια ο αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής ο κύριος όλι θα ήθελε να κάνει μια δήλωση. Πολύ θα ήθελα να είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. τα πυροτεχνικά είδη βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια κυρία Ρόιτοβα για τις εργασίες της, για την πρόταση που μας έκανε σε πνεύμα συμβιβασμού και για να καταλήξουμε σε συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση, η Επιτροπή δεν θα παρεμποδίσει αυτή τη συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και γι' αυτό καλωσορίζουμε αυτό το πακέτο συμβιβασμών και προσβλέπουμε στην σύντομη έγκριση του. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής που δημιουργεί αυτή η οδηγία και έχει στείλει μια δήλωση ε, προς το Κοινοβούλιο ε, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία επί της ε, έκθεσης του κυρίου Μπόρη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Εξετάζουμε την πρόταση ψηφίσματος. Παράγραφος 5 σε δύο τμήματα ε, πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 28 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση έναρξη της ψηφοφορίας λήξη Εγκρίνεται. Παράγραφος 29 ε, με ονομαστική κλίση, έναρξη, λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 30 με ονομαστική κλίση, έναρξη, λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 42 με χωριστή ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 44 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 45 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 47 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 54 με ονομαστική κλίση έναρξη της ψηφοφορίας Λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 69 με χωριστή ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέτω το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται Συγχαρητήρια στον κύριο Μπόρις. Καλή σας όρεξη. So uh, apparently there was an agreement between